19 Μαΐου 12 το μεσημέρι. Η δε Τετάρτη 20 Μαΐου. Η κυρία Πίρκο Ρούχονεν Λέρνερ αντικαθιστά τον κύριο Σαν ως Ευρωβουλευτής, ως μέλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από 27 Απριλίου 2015. Ε, μας ενημερώνουν οι φιλανδικές αρχές, την καλωσορίζουμε και